Pan So good afternoon, colleagues. We can start our... Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε τα πρακτικά της χρησινής συνεδριάσεως, τα έχετε στην κατοχή σας, εάν δεν έχετε ενστάσεις θεωρώ ότι εγκρίνονται. Το επόμενο, και, επόμενο θέμα δηλαδή και πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζητήση περιπτώσεων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Πρώτο θέμα, Πακιστάν, δολοφονία του κυβερνήτου της επαρχίας του Πουντζάμπ, Σαλμάν Τασέρ. Το λόγο θα δώσω πρώτα στους συντάκτες την κυρία Σάκερ δηλαδή, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε Φίλε, συνάδελφοι. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος αγώνας που δίνεται στο Πακιστάν. Ε, τα τάσεις που έχουμε δει, οι εξτρεμιστικές τάσεις πρέπει να πάυσουν. Είδαμε ότι δημιουργείται ένα κλίμα φόβου και ε, έλλειψης ανοχής και εξτρεμιστικών τάσεων. Αυτό δεν είναι απλό καθήκον για μας να αντιμετωπίσουμε τον εξτρεμισμό. Και για το Πακιστάν και για όλους τους πολίτες που συμφωνούν ότι η μη ανοχή και ο φόβος πρέπει να πάυσουν. Πρέπει να εκριζώσουμε την τρομοκρατία. Ο κυβερνήτης ε, Τασίρ δολοφονήθηκε άγρια ακριβώς για λόγους μη ενοχής από ένα ίδιο μέλος της ε, φρουράς του. Από ένα μέλος της ίδιας του φρουράς μάλλον. Η κόρη του έγραψε μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στις New York Times και θα ήθελα να παραθέσω ένα μέρος της επιστολής της γιατί νομίζω ότι λέει τα πράγματα με πολύ, περιγράφει τα πράγματα με πολύ σωστό τρόπο. Και σε μνήμη του πατέρα της θέλω να θυμίσω όσα λέει. Μιλά για το δράστη λοιπόν. Λέει ότι ο δράστης και οι υποστηρικτές του επέφεραν ένα βαρύ πλήγμα εκείνη τη μέρα αλλά ότι ε, έχουν μεγάλε αυταπάτε αν πιστεύουν ότι θα θυμώσουν τη φωνή του πατέρα τη και πολλών άλλων χιλιάδων πολιτών του Πακιστάν που πιστεύουν ε, στην ε, ελευθερία στο Πακιστάν. Επίση, υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι ο πατέρα, ο θάνατο του πατέρα μου, ε, δείχνει το τέλο τη ανοχή στο Πακιστάν και ότι επιπλέον οι φωνέ υπέρ τη ελευθερία στο Πακιστάν θα πάυσουν. Όχι, αυτή η θαραλέα φωνή θα εμπνεύσει και άλλους. Άλλοι, άλλοι ακολούθησαν την και αντέδρασαν στην ε, έγκριση του νόμου για τη βλασφημία, ε, ιδίω ακόμη και συντηρητική πολιτική. Και να θυμίσω ότι η κόρη του κυρίου Τασίρ πήγε στο, Σμίθ, στο κολέγιο Σμιθ και ε, μελέτησε Ευρωπαϊκό Δίκαιο και για ανθρώπινα δικαιώματα. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η νέα γενιά στο Πακιστάν πρέπει να έχει ευκαιρίε και δικαιώματα και τη δυνατότητα να ζει σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπω αυτή του Πακιστάν. Ευχαριστούμε ο κύριος Είδαμε το τι έγινε στο Πακιστάν και είδαμε το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση στη χώρα. Ο κύριος Τασεέρ ήταν ο κυβερνήτης της μεγαλύτερης επαρχίας της χώρας και πέθανε γιατί ήταν θαραλέος γιατί είχε το θάρρος ε, να υπερασπίσει τους χριστιανούς και να υπερασπίσει ε, μια καταδικασμένη σε θάνατο. Πρόκειται για ε, κάποιον ο οποίος δεν φοβήθηκε να μπει στο στόχαστρο των φανατικών Ισλαμιστών. Βλέπουμε πως οι πολιτικές ελίτ, πως το δικαστικό σύστημα έχουν υποκύψει σε τεράστιες απειλές, τις απειλές των Ισλαμιστών. Εμείς ε, ε, ψηφίσαμε για την προστασία των χριστιανών. Ε, θα ήθελα η κυρία Άστον να ασκήσει πιέσει στο Πακιστάν για, για την πράστηση των χριστιανών. Η κυρία Κορόλα, ένα λεπτό. Δεν ήταν έκπληξη πραγματικά όταν λάβαμε τα νέα ότι δολοφονήθηκε ο, ο κυβερνήτης ε, Σαλμαν ήδη την κυρία Μπούτο και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του Πακιστάν. Γνωρίζω και την περίπτωση της ε, καταδίκης και της δίωξης μάλλον για λόγους βλασιμίας. Η πακιστανική κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικά βήματα για να βελτιώσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων, δίνοντας για παράδειγμα ποσοστώσεις σε δημόσιες θέσεις. Πρέπει όμως να επανεξετάσει όλους τους νόμους που οδηγούν σε διακρίσεις μεταξύ αυτών και τον νόμο κατά της βλασφημίας. Χρειάζεται να ελευθούν και άλλα μέτρα γιατί εξακολουθούν και υπάρχουν μεγάλα κενά όπως για παράδειγμα στον παρόντα νόμο περί βλασφημίας που επιτρέπει στους σε ακραίους, σε εξτρεμιστές να λαμβάνουν δράση. Ελπίζω ότι με το ψήφισμά μας θα μπορέσουμε να εκφράσουμε τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μας με την κυβέρνηση του Πακιστάν στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας και κατά της ανάπτυξης του εξτρεμισμού. Ευχαριστώ κύριε Κορχόλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από 8 μήνες, στις 20 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα για την ελευθερία ε, θρησκεύματος ε, στο Πακιστάν. Σήμερα το ίδιο θέμα βρίσκεται εδώ στο σώμα μετά από την καταδίκη σε θάνατο της κυρίας Σαμπίμπη και της δολοφονίας του αυτού που την υπερασπίστηκε δημόσια. Σήμερα το Πακιστάν κάποιος μπορεί να θανατωθεί για βλασφημία, για την έλλειψη ε, ε, ε, ελευθερίας του λόγου. Βλέπετε λοιπόν πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση μπροστά μας. Δολοφονούνται οι τοπικές ελίτες σε αυτή τη χώρα όπου είναι μισοί χριστιανοί και οι μισοί Ισλαμιστές. Το άρθρο 5 του Πακιστανικού Συντάγματος μπορεί να καταδικάσει σε θάνατο κάποιον για βλασφημία. Πρέπει να υποστηρίξουμε το Υπουργείο Μειονοτήτων ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται στην για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα στην οποία αντιστέκεται η Ισλαμική Λίγα. Θα πρέπει να καταργηθεί λοιπόν αυτό το άρθρο και να ισχύσει το Σύνταγμα του 73 για την ανεξιθρησκεία. Η κυρία Βεργιά για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ ε, θα ήθελα να πω ότι διάβασα το κοινό ψήφισμα ε, στο, για το Πακιστάν και τη δολοφονία του κυβερνήτη Ταζέρα με ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μιλήσαμε σήμερα για τις χριστιανικές μειονότητες. Όλοι μας είμαστε συνδεδεμένοι με την ελευθερία της συνείδησης και θρησκείας και θα πρέπει να ανησυχούμε για όλους όσους διώκονται για τις επιλογές τους, τις θρησκευτικέ τους επιλογές όταν αλλάζουν θρησκεία ή όταν δεν πιστεύουν στο Θεό. Αν εμείς θέλουμε να παλέψουμε κατά του θρησκευτικού ολοκληρωτισμού θα πρέπει να βοηθήσουμε όλους και όλες είναι θύματα αυτού του φανατισμού. Καμία θρησκεία δεν, ε, δεν είναι άμεμπτη. Θυμηθείτε τις μαζικές δολοφονίες των ε, ε, Ινδιάνων στην Αμερική ή των σκλάβων στην Καρυβική. Θυμηθείτε τους ε, θρησκευτικούς πολέμους, ε, θυμηθείτε τον, αντισημιτισμό ο οποίος βιώνει σε λανθάνουσα μορφή σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φανατική ε, είναι υπεύθυνοι αλλά και οι μετριοπαθείς ε, που τους, ε, που τους καλύπτουν πληρώνουν επίσης. Αυτός ο άνθρωπος στο Πακιστάν, ο κυβερνήτης, καταδίκασε τον νόμο για τη βλασφημία στη χώρα του και για το πώς χρησιμοποιούσαν αυτόν τον νόμο οι εξτρεμιστές εναντίον ας πούμε της γυναίκας η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο για βλασφημία. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο νόμος για τη βλασφημία εφαρμόζεται πρώτα απ' όλα κατά των μουσουλμάνων. Το ότι πλήττει όλες τις θρησκευτικέ μειονότητες, κυρίως τις γυναίκες, τους συνδικαλιστές, τους δικηγόρους και αυτοί οι άνθρωποι στερούνται των θεμελιωδών τους ελευθεριών ή αναγκάζονται να ζήσουν σε παρανομία. Θα ήταν λοιπόν καιρός η Κομισιόν και οι υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων να αλλάξουν τις πολιτικές τους και θα ήθελα κύριε Επίτροπε να μας κάνετε έναν απολογισμό συγκεκριμένο για τη συμφωνία με την Τινησία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης στο Πακιστάν. Η Τινησία να μας γίνει μάθημα ολονών και σας. Η κυρία Λαμπέρτ για δύο λεπτά. Νομίζω όλοι εδώ θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μα στην οικογένεια και του φίλου του Σαλμάν Ταζίρ, του κυβερνήτη του Πουντζάμπ. Το τίμημα Βεβαίω θα το πληρώσει η κυβέρνηση του Πακιστάν. Ε, και εδώ να θυμηθούμε τη σαφή του στήριξη, καθώ ε, όντα την αντιπολίτευση ήξερε να υψώνει τη φωνή του και μπορούσε να γίνει και επικίνδυνο. Νομίζω δικαίω λοιπόν να θλιβόμαστε όλοι για τη δολοφονία του και ε, παίρνουμε το μέρο του πληθυσμού του Πακιστάν που καταδικάζει αυτή τη δολοφονία. Όμω δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι κι άλλοι τον θρύνησαν και κάποιοι δημοσίω. Αυτό είναι μια δημόσια πράξη. Άρα θα πρέπει να επενέσουμε και τη δράση του ρυθμιστή μάλλον να καταδικάσουμε τη δράση του ρυθμιστή των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης, του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, που ε, απαγόρευσε δημοσιεύματα που έδιναν στοιχεία για τον ε, δράστη, τον ύποπτο για την δολοφονία. Πάντως, στην κοινωνία του Πακιστάν υπάρχουν πολλές διαφορετικές, πολλά διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα, χριστιανικό, ε, μουσουλμανικό και ούτω καθεξής. Το Πακιστάν είναι μια νέα δημοκρατία που αντιμετωπίζει πιέσεις στα σύνορά του, αντιμετωπίζει φυσικές καταστροφές ε, λόγω των πλημμυρών και τον σεισμό της περασμένης εβδομάδας. Αλλά δίνει τη μάχη του και αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται τη στήριξή μας στο Πακιστάν προκειμένου να αναπτυχθεί το δημοκρατικό καθεστώς αυτή τη χώρα. Όχι ε, μόνο για να αντιμετωπιστεί ο εξτρεμισμός και να προστατευτούν καθολικοί κόστα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά γιατί και οι δημοκρατικά εκλεγμένοι βουλευτέ θα πρέπει να ε, ε, στηριχθούν και όλοι εμεί ε, ω ομόλογοι του εκτό Πακιστάν να του βοηθήσουμε να ακουστεί η φωνή που προσπαθούν να φημώσουν. Ακούσαμε την πρόσφατη δράση τη κυβέρνηση του Πακιστάν. Θα πρέπει να αρθούν οι ενδιασμοί του διεθνούς ε, απαγορευτής, διεθνής απόφασης ε, για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών δικαιωμάτων που πρόσφατα εγκρίθηκε. Αυτά τα είπαμε και σε πρόσφατη επίσκεψή μας στο Πακιστάν με την αντιπροσωπεία μας. Πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα να τροποποιηθεί ο νόμο κατά τη βλασφημία. Διότι ο νόμο αυτό είναι καταχρηστικό. Και περισσότερο γίνεται καταχρηστή του παρά χρήση του. Τώρα θα ακολουθήσουν οι αγορητέ των πολιτικών ομάδων και ο πρώτο ο κύριο Κέλαμ για ένα λεπτό εξ ονόματο του Λαϊκού κόμματο. Όλοι καταδικάζουμε αυστηρά την ε, δολοφονία του κυβερνήτου του Πουντζάμπου στις 4 Ιανουαρίου. Ο φόνος αυτός διεξήχθη διότι ο Τασίρ αντιτάχθηκε στον διαβόητο νόμο περί βλασφημίας που επιτρέπει καταπίεση άλλων θρησκευτικών ομάδων. Με την έκφραση ανησυχίας λόγω της αυξανόμενης, της αυξανόμενης επιρροής των εξτρεμιστών στο Πακιστάν, στο Πακιστάν οφείλουμε να κατανοήσουμε ωστόσο και οι μετριοπαθείς της κυβέρνησης του Πακιστάν, μεταξύ των οποίων συγκατελέγεται και ο κ. Στασίρ, υπέστησαν σοβαρή απώλεια και θα πρέπει να τους συλληπιθούμε. Ανησυχούμε για το γεγονός ότι νεαροί δικηγόροι επένεσαν τον δολοφόνο. Ωστόσο, στο μεγάλο, μεγάλο μέρος της κοινωνίας του Πακιστάν καταδίκασε τον φόνο. Ακόμη και θρησκευτικέ αρχές ζήτησαν τροποποίηση του νόμου περιβλασιομίας και συμπαρατασσόμαστε στην αξίωσή τους αυτή. Σας ευχαριστώ. Mr. Kellam, now on behalf... Ευχαριστώ κύριε Κέλαμ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ κυβερνήτης του Πουντζάμπ, Σαλμάν Τασίρ, δολοφονήθηκε σε μια εκδήλωση θρησκευτικής δυσανεξίας από μέρος της κυβέρνησης από μέρος συγγνώμη, της, ε, της κοινωνίας του Πακιστάν. Είχε ζητήσει την απόλυση από τις φυλακές της χριστιανής Μπινίν. Ποια είναι η μοίρα ανθρώπων που ε, υφίστανται τέτοιε διώξει. Δηλαδή, εάν απολυθεί τελικά από τι φυλακέ η Μπινίν, κινδυνεύει και αυτή να δολοφονηθεί. Υπάρχει έλλειμμα προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων στην χώρα αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Ρέπο. Εκ μέρου των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, η κυρία Όγιουλαν. Για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η δολοφονία του κυβερνητή Σαλμάν Τασίρ δεν είναι μόνο μια ιδιωτική τραγωδία, προσωπική τραγωδία της οικογένειάς του, αλλά μια δημόσια τραγωδία για την δημοκρατία στο Πακιστάν. Παρόμοιες περιπτώσεις που αναφέρονται στο ψήφισμά μας, όλες μαζί, δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση εκφοβισμού από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κοινωνία του Πακιστάν, ώστε να υπάρξει τάση ριζοστική προσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού θρησκευτικού στη χώρα ε, να επιταθούν τα φαινόμενα αυτά. Και ε, ο νόμος ε, κατά της βλασφημίας δεν συνάδει με το σύνταγμα της χώρας. Ε, έτσι δημιουργήθηκε το κλίμα αυτό που οδήγησε στην δολοφονία του Σαλβάν Τασίρ. Πρέπει να σκεφτούμε τις διακλαδώσεις και τις συνέπειες της εφαρμογής τέτοιων απάνθρωπων νόμων σε ευαίσθητες κοινωνίες όπως αυτή του Πακιστάν. Το Πακιστάν θα επωφελεί το κατά πολλού τρόπους αν ανακαλούσε το νόμο αυτό κατά της βλασφημίας και τι ποινέ που επιβλήθηκαν βάσει του νόμου αυτού. Ελπίζουμε η κυβέρνηση του Πακιστάν να ενισχύσει τα μέτρα που ε, είχε εγκρίνει ώστε να καταπολεμήσει την εξάπλωση του βίαιου εξτρεμισμού. Ο εξτρεμισμό οδηγεί σε βία και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη Μάλλον είμαι απόλυτα βέβαιη ότι το Πακιστάν δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την κλιμάκωση ενό ε, διευρυμένου εμφύλιου πολέμου, όπου θα συμμετείχαν ενδεχομένω και τα Λιμπάν. Ευχαριστούμε και τώρα από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, ο κύριο Τσανέσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάλι μιλάμε για το Πακιστάν και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή και βλέπουμε να εξετάζουμε μια πολιτική εδώ δολοφονία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ε, συζητούμε τέτοια θέματα. Εγκρίναμε ψηφίσματα, ένα ψήφισμα πριν από λίγους μήνες για το Πακιστάν και πάλι και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που είναι αντί να αντιμετωπιστεί. Ε, Εδώ μιλάμε για προβλήματα ανεκτικότητας, μυσαλλοδοξίας. Μιλάμε για τους μουσουλμάνους ημάμιδες, οι οποίοι δημοσίως εκδηλώνουν τη μυσαλλοδοξία τους στο Πακιστάν τάσσονται υπέρ της δολοφονία, των δολοφονίων σαν αυτές που αναφέραμε και προσφέρουν και ε, επικηρύξεις ε, και αμοιβέ για τέτοιου είδους δολοφονίες. Η κυβέρνηση του Πακιστάν δεν αντέδρασε επισήμως. Θα πρέπει λοιπόν να... Είμαστε ε, σαφείς. Η αδράνεια είναι υπεύθυνη για τη βία. της ομάδας Ευρώπη για τη Δημοκρατία, ο υποκόμις του Dartmouth για να μπορέσω να κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Όταν ήμασταν 20 και περισσότερο ετών, ήμασταν φίλοι με τον Σαλμάν Τασίρ και με, μου έγραψε στο κοινοβούριο ο Σαλμάν και με προσκάλεσε ως ιδιωτικό του προσκεκλημένο στο Μέγαρο ε, στην, κυβέρνηση στο Πακιστάν. Αυτή η επιστολή έφτασε σε μένα μετά την δολοφονία του. Ο Σαλμάν ήταν άνθρωπος με χάρισμα ταλέντο και υψηλότατη ευφυΐα. Άνθρωπος επίσης αποτελεσματικός. Εκπροσωπούσε τις καλύτερες παραδόσεις του Πακιστάν. Μουσουλμάνος αλλά κατ' ουδένα τρόπο φανατικός. Υποστήριξε μια χριστιανή η οποία καταδικάστηκε υπό την ισχύ του νόμου περιβλασιμίας και αυτή την υποστήριξη την πλήρωσε με την ζωή του. Επρόκειτο για πολιτική δολοφονία. Το Πακιστάν δεν είναι μονάχα μια μεγάλη αναπτυσσόμενη χώρα, είναι μια χώρα η οποία έχει και πάνω από 20 πυρηνικέ κεφαλές. Προσήλθα εδώ σήμερα πρώτα για να εκφράσω την μεγάλη προσωπική βαθιά μου θλίψη για το γεγονός αυτό, αλλά ταυτόχρονα και τι ανησυχίε μου και τι ανησυχίε όλων μα για την πορεία του Πακιστάν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε, ο κύριος Μαν ακολουθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο βίο θάνατο του κυβερνήτου του Πουντζάμπ Σαλμάν Τασίρ που ήταν πάντοτε υπέρ μιας ανεξιθρησκείας τρόμαξε όλο τον κόσμο. Δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν, όχι όμως κατά του φόνου, αλλά υπέρ του δολοφόνου. Ο Τασίρ ήταν αντίθετο με τον νόμο περί βλασφημίας, ο οποίος επιβάλλει ποινή θανάτου σε περιπτώσεις βλασφημίας του θείου στο Πακιστάν. Οι χριστιανοί Μπιμπίν καταδικάστηκε πρόσφατα σε θάνατο για δίθεν προσβολή του προφήτου Μωάμεθ. Το Λαϊκό Κόμμα έχει ταχθεί πάντοτε κατά, της, ε, κατά του εξτρεμισμού. Ο θάνατος του Σαλμάν Τασίρ ε, αποτελεί μεγάλο σημάδι. Υπάρχει περίπου ένα εκατομμύριο χριστιανών. Τι θα υποστούν αυτοί ακόμη. Η Ευρώπη οφείλει να αναμειχθεί και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Νότιο-Ανατολική Ασία, της οποίας είμαι αντιπρόεδρος, πρέπει να θέσει το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει να υπάρξει διαρεύνηση του φόνου. Πρέπει να αχθούν ενώπιον των δικαστηρίων και να υποστούν τις συνέπειες ο δολοφόνος του και οι υποστηρικτές του. Ο κ. Παλέτσκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Πακιστάν αρχίζει να γίνεται έκρηθμη. Ε, λόγω και των εξωτερικών και των εσωτερικών ε, συνθήκων ε, των πολιτικών. Άρα τέτοια γεγονότα όπως ε, μια πολιτική δολοφονία λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων μιας γνωστής προσωπικότητας κλονίζουν ολόκληρη τη χώρα και την κοινωνία της. Οι συνέπειες από τέτοια γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης στη χώρα δεν θέλουμε να, ξέρετε, να ε, επιτείνεται ο θρησκευτικό φανατισμό στην ε, χώρα αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε την εξή πορεία. Αυτό το υποδεικνύει και το ψήφισμά μα. Να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα γεγονότα να πάρουν μια άλλη τροπή. Να επηρεάσουμε την κυβέρνηση του Πακιστάν ώστε να αναζητήσει ε, δυνάμει στη χώρα και να αντισταθεί στην έλλειψη θρησκευτική ανοχή και ανεκτικότητα. Θα πρέπει λοιπόν μια τέτοια πορεία να την υποστηρίξουμε ενεργά και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Διότι έχουν πολλέ φορέ να εκδικάσουν πολύ δύσκολε υποθέσει, ιδίω αυτέ που βασίζονται στο νόμο περί πλασφημία. Και τώρα ο κύριο Σόγκορ Τσάμπα. E Ήδη κατ' επανάληψη έχουμε τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταδικάζει τις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Ευρώπη δεν επιτρέπεται να αφήσει στη μοίρα τους ανθρώπους οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ίσης μεταχείρισης των μειονοτήτων. Γνωρίζουμε ότι διώκονται χριστιανοί σε πολλές χώρες και όχι μόνο στο Πακιστάν. όχι μόνο, δεν χρειάζονται μόνο στο Πακιστάν ηγετικέ προσωπικότητες όπω ο Σαλμάν Τασίρ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω πρέπει να δώσει σάρκα και οστά στι ευρωπαϊκέ αξίε. Η ανεξιθρησκεία είναι κοινή μα αξία και μπορούμε να λαμβάνουμε εαυτού σοβαρά μονάχα εφόσον προσφέρουμε την υποστήριξή μα στους Χριστιανού και στι άλλε θρησκευτικέ μειονότητε. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στη διαδικασία Catch the Eye, προσέλκυση της προσοχής. Έχω βέβαια 14 συγγεγραμμένου ήδη. Όλοι θα λάβετε χρόνο σα, αλλά περιοριστείτε απολύτω και αυστηρό σε ένα λεπτό. Ο κ. Σιλβέστρης. Κύριε Επίτροπε, δεν μπορεί να μένει άπραγη η Ευρώπη μπροστά σε αυτό το οποίο συμβαίνει στο Πακιστάν. Η δολοφονία του κυβερνήτη του Ποντζάμπ είναι πάρα πολύ σοβαρή. Η κατάσταση χειροτέρεψε αυτούς τους μήνες. Η διαμάχη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων είναι πάρα πολύ σοβαρή αλλά οξύνθηκε με την νομοθεσία για τη βλασφημία και ο κυβερνήτης του Πεντζάμπ εξέφρασε την ε, διαφωνία τη με, αυτή την καταδίκη και γι' αυτό δολοφονήθηκε. Είναι ένας μετριοπαθής, γι' αυτό λοιπόν και δολοφονήθηκε. η έλλειψη μιας ισχυρής παρέμβασης εκ μέρους της Ευρώπης θα οδηγούσε στην όξυση των εξτρεμιστών. Ευχαριστώ που κρατήσατε το χρόνο σας, ο κύριος Αρλάκη. Πρόεδρε, πέραν των επικρίσεων, ένα μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινού και μέρος των βουλευτών μας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 έχουν αμφιβολίε για τον αγώνα του Πακιστάν κατά τη τρομοκρατία. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια του Πακιστάν και βλέπω και τι προσπάθειε τη κυβέρνηση του Πακιστάν και τη κοινωνία των πολιτών κατά των εκτρεμιστών. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί προ όλου. Το 90% και περισσότερο του λαού του Πακιστάν είναι κατά τη τρομοκρατία και πληρώνουν ένα πολύ βαρύ τίμημα για τι τρομοκρατικέ ενέργειε στη χώρα του. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι ο κύριο ε, Τασίρ Τη δολοφονία του μάλλον την καταδίκασε η πλειοψηφία του λαού του Πακιστάν, καθώς και μέλη επίσημα της κυβέρνησης. Ε, οι, μουσουλμαν, οι εκπρόσωποι ε, του μουσουλμανικού χώρου και πολλά μέλη της κυβέρνησης εξέφρασαν τη θλίψη τους για το γεγονός αυτό. Θα πρέπει αυτό να αναγνωριστεί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ελευθερία θρησκευτικής έκφρασης είναι από τα πλέον θεμελιώδη δικαιώματα και όμως παραβιάζεται καθημερινά σε διάφορα τμήματα του κόσμου. Αυτό είναι βαρύτατη ε, παραβίαση. Τα όσα συνέβησαν στο Πακιστάν έχουν σχέση και με την παλαιότερη στρατιωτική δικτατορία που κατά λοιπά επιμένουν να ε, καταπιέζουν τις μειονότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει ώστε η πακιστανική κυβέρνηση να αποσύρει τον βάρβαρο αυτόν νόμο. Τσάρλ Στάνοκ. Όταν ετάφη ο κυβερνήτης Τασίρ μου φάνηκε ότι ετάφη μαζί του και κάθε ελπίδα για πρόοδο στο Πακιστάν πρέπει να τροποποιηθεί αυτός ο δρακόντιος νόμος περί βλασφημίας και να απολυθεί η χριστιανή η οποία να μένει εκτέλεση θανατικής ε, ποινή για δίθεν βλασφημία κατά του προφήτου. Χρειάζεται υποστήριξη από πλευρά μας των θρησκευτικών μειονιτήτων. Προχωρεί η ριζοσπαστικοποίηση της ε, ε, πακιστανικής κοινωνίας. Ελάχιστοι πολιτικοί στο Πακιστάν τολμούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Τασέρ και μάλιστα ακόμα λιγότερο τώρα όπου θα φοβούνται. Δυστυχώς οι φανατικοί μεταξύ αυτών και σημαντικοί νομομαθείς στο Πακιστάν επενούν τον δολοφόνο και φαίνεται να κερδίζουν τον πόλεμο ιδεών στο Πακιστάν. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει στρατηγική σχέση και μάλιστα με τις γενναιότερες αυτές παραχωρήσεις ε, στο εμπόριο. Σας ευχαριστώ, κ. Σκέλη. Εδώ μιλάμε για μια φρικτή τραγωδία. Πρώτα απ' όλα για την εκτέλεση ενός αθώου ανθρώπου και έπειτα για την εκτέλεσή του από έναν από τους δικούς του ανθρώπους της φρουράς του, το σωματοφύλακά του. Εδώ πρέπει να θυμίσω ότι μόλις πριν από μια εβδομάδα είχα μια παρόμοια εμπειρία διαφορετικές διαφορετικές συνθήκες. Βρισκόμασταν Μάλλον βρισκόταν ένα εκπρόσωπο της Ιρλανδίας ε, στον Άγιο Μαυρίκαιο για το μήνα του μέλητο και δολοφονήθηκε από μέλος της φρουρά του στην κρεβατοκάμαρα του ξενοδοχείου. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ένας αθώος χάνει τη ζωή του για πολιτικούς λόγους. Ήμουν μέλος της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας ε, για το Πακιστάν και είχα συναντήσει τον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος μου μίλησε με πολύ λογικό τρόπο και με σταθερό τόνο και μου είπε ότι θέλει να εμποδίσει την έξαρση του θρησκευτικού εξτρεμισμού στη χώρα. Ε, θα τους αντιμετωπίσει όπως μπορούσε, μου είχε πει. Γνωρίζουμε τις προσπάθειες της χώρας αυτής. Ε, ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η δολοφονία του κυρίου Τασίρ έχει ένα ιδιαίτερο νόημα λόγω του τοπίου στο οποίο έλαβε χώρα του πολιτικού σκηνικού. Φαίνεται να υπήρχε μια μυστική έγκριση τη δολοφονία αυτή από του πνευματικού ηγέτε του Πακιστάν. Τι σημαίνει αυτό, Ότι οι δολοφονίε και οι φόνοι είναι μέσα που επιτρέπονται πλέον από του θρησκευτικού ηγέτε του Πακιστάν και μάλιστα παροτρύνονται. Ε, ο νόμος κατά της βλασφημίας τιμωρεί απλούς ανθρώπους με ποινές όπως και τη θανατική καταδίκη και οδηγεί στην απώλεια ζώων. Πρέπει λοιπόν εδώ να, να αντισταθούμε. Θα πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση του Πακιστάν να αλλάξει αυτή την κατάσταση και άλλες κυβερνήσεις να ασκήσουν και εκείνες πιέσεις. Δεν μπορούμε να αποδειχόμαστε στον 21ο αιώνα να συμβαίνει κάτι παρόμοιο και να γυρνάμε στο μεσαίωνα. Ευχαριστούμε ο κύριος Σακέντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πρώτον η κατάσταση στο Πακιστάν είναι ανησυχητική γενικά και όχι μόνο λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το Πακιστάν είναι μακριά μας γιατί γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που σημειώνονται εκεί είτε είναι οικονομικά είτε είναι μεταξύ μειονοτήτων είτε είναι πολιτικού χαρακτήρα έχουν σημαντική επιρροή διότι προκαλούν μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα καλούμαστε να αναλάβουμε δράση. Υπάρχουν δύο προβλήματα που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Αφενός, οι συνεχείς επιθέσεις από, από Αφγανιστάν και από Ινδία, προς το Πακιστάν δηλαδή, και επίσης οι μουσουλμάνοι εξτρεμιστές οι οποίοι δολοφόνησαν τον κυβερνήτη Τασίρ. Γι' αυτό ζητώ από το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει το Πακιστάν στην διερεύνηση της υποθέσεως. Η κυρία Μακοβέη. Η δολοφονία του κυβερνήτη του Πουντζάμπ μια από τι φωνέ που υποστήριζε την ανεκτικότητα και την προστασία των μειονοτήτων στο Πακιστάν δείχνει την ε, δραματική αύξηση των περιπτώσεων παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Η θύμωση τη ελευθερία έκφραση, η η έκφραση των θρησκευτικών επιθήσεων τιμωρείται με φυλάκιση και η κάθερξη ή και θανατική καταδίκη. Ο κύριο ε, Τασίρ έχασε την ελευθερία του και μετά και τη ζωή του γιατί υποστήριζε την ελευθερία των υπολείπων. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίζουμε όσου είναι τελμηροί να υποστηρίζουν τέτοιου είδου ε, αξίε όπω την δημοκρατία και την ελευθερία. Εδώ θα πρέπει να παροτρύνουμε τι ε, πακιστανικέ αρχέ να τιμωρήσουν τους του δράστε, του υπευθύνου, όσου είναι εξτρεμιστέ και να, να ανακλάλουν, αλλά καλέσουν τον νόμο κατά τη βλασφημία. Uh, Πρόεδρε, η δολοφονία του κυβερνήτη Τασίρ είναι ένα φρικτό και αποτρόπαιο έγκλημα. Ε, φαίνεται ότι ο δράστη ήταν ένα εξτρεμιστή, γιατί εκείνο πρότεινε τροπολογίε, ε, ο κυβερνήτης πρότεινε τροπολογίε στον νόμο κατά τη βλασφημία. Τι σημαίνει τώρα η κατάσταση του Πακιστάν για τη Δύση. Σημαίνει ότι αντί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, κατα... για να αναχαιτήσουμε τον ε, μουσουλμανικό εξτρεμισμό και την εξάπλωσή του στην Ευρώπη, τελικά προσπαθούμε να χαλαρώσουμε απλώ την αντιμετώπιση του. Εδώ βλέπουμε τον νόμο για την Σαρία στην... στον Βασίλειο και Βλέπουμε ήδη τέτοιες περιπτώσεις γύρω μας. Εδώ είχαμε το διαφωτισμό, την βιομηχανική επανάσταση, τα, θαύματα του σύγχρονου επιστημονικού κόσμου. Δεν μπορούμε να περνάμε σε, ιδεολογικά, σε ιδεολογίες και πιστεύω πριν από τον 6ο αιώνα. Ε, εδώ χρειάζεται να είμαστε πολιτικώς λογικοί και να αναχαιτήσουμε την ε, πολιτική ισχύ των ε, εξτρεμιστών στις μουσουλμανικές χώρες, να στηρίξουμε τις προοδευτικές δυνάμεις στο Πακιστάν και να βεβαιωθούμε ότι ο νόμος για τη Σαρία και ο ο εξτρεμισμός των Ισλαμιστών δεν θα ριζώσει και στις δυτικές δημοκρατίες. Ευχαριστούμε ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, επιθυμώ να πω ότι καταδικάζω την βάρβαρη δολοφονία του κυβερνήτη του Πουντζάμπ. Σημαντική προσωπικότητα της δημόσιας ζωής του Πακιστάν που κατέστη γνωστός για τον αγώνα του κατά του φανατισμού. Προμηνών είχαμε μιλήσει για την ανάγκη αγώνα κατά του νόμου της περί βλασφημίας. Υπενθυμίζω ότι οι καταχρήσεις του που επιτρέπει ο νόμος αυτός οδηγούν σε μεγαλύτερη έλλειψη ανοχής απέναντι σε θρησκευτικές μειονότητες καθώς επίσης και σε διακρίσεις. Στην περίπτωση της Άσια Μπίμπη που τελικά προκάλεσε και την δολοφονία του κυβερνήτη Τασέρ αποτελεί ένα παράδειγμα. Πρέπει να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει σημασία στον αγώνα κατά του εξτρεμισμού στη χώρα αυτή. Απευθύνω έκκληση στις φωνές της λογικής στη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, Μικολάσικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στους πολίτες του Πακιστάν που έχασαν μια σημαντική ηγετική προσωπικότητα τον κυβερνήτη Σαλμάν Τασέρ. Με ανησυχεί το γεγονός ότι άνθρωποι στη χώρα αυτή διώκονται επειδή έχουν διαφορετικές θρησκευτικέ πεπιθήσεις και δεν αποτελούν εξαίρεση θρησκευτικές θρησκευτικέ ομάδες όπως οι χριστιανοί. Μια γυναίκα η οποία καταδικάστηκε στη βάση του νόμου της Σαρίας έχει καταδικαστεί σε θάνατο Το πρόβλημα είναι ότι οι δυνάμεις δημοσίας τάξεως και ασφάλειας στο Πακιστάν αριθμούν εξών των μελών τους πάρα πολλούς μουσουλμάνους φανατικούς. Θα ζητήσω από όλες τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και από τις θρησκευτικές αρχές να υποστηρίξουν τις μετριοπαθείς φωνές μεταξύ των κοινοτήτων. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι έφραστη χώρα το Πακιστάν από πολλές απόψεις και διότι η κυβέρνηση δεν είναι ικανή να τηρήσει και να επιβάλλει την μετριοπαθή στάση που επιθυμεί, ο στρατός διότι αντιμετωπίζει στα σύνορα του Πακιστάν ε, επίμονες επιθέσεις των εξτρεμιστών η οικονομία είναι έθραυτη αλλά και κοινωνικά είναι έθραυτη η χώρα αυτή διότι επί δεκαετίε η κοινωνία δεν αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο που να επιτρέψει συμμετοχή μεγάλων τμήματων τη κοινωνία σε μια οικονομική ανάπτυξη. Ω Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογό μα με την πολιτική τάξη και να προωθήσουμε την αντίληψη ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι προσπάθειες για οικονομική ανάπτυξη, ώστε να καταδειχθεί στους ανθρώπους εκεί ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες να βελτιώσουν τη ζωή τους και όχι μόνο με τον θρησκευτικό φανατισμό. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Τελευταίος είναι ο κύριος Πόσελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πλέον εμοσταγή καθεστώτα ήταν τα ε, αντιθρησκευτικά καθεστώτα των Ιακωβίνων, των Εθνικοσοσιαλιστών και των Κομμουνιστών στην Ευρώπη. Δεν συμβάλλει όμως η κυρία Βεργιά όταν στρέφεται κατά των θρησκειών συνολικά. Συχνά τις θρησκείες τις εκμεταλλεύονται ορισμένοι για λόγους πρόθεσης φανατικών ιδεών. Το Πακιστάν όμως προέκυψε από τον χωρισμό της Ινδίας μετά από την ε, Βρετανική ε, την αποχώρηση από εκεί για λόγους θρησκευτικού για να έχουν χώρο οι μουσουλμάνοι. Ωστόσο η χώρα αυτή οφείλει να σεβαστεί τις θρησκευτικές πεπιθήσεις των υπολείπων ομάδων και τους χριστιανούς ιδιαίτερα, υπέρ των οποίων θα πρέπει να παρέμβουμε εμείς πολύ πιο ενεργά από ό,τι το πράξαμε μέχρι τώρα. Διότι ποιος θα υποστηρίξει τους χριστιανούς ανά τον κόσμο, αν όχι εμείς οι Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ και πώς Βλέπω και την κυρία Εσάγια που θα είναι αυτή πραγματικά η τελευταία μας ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πολλοί είναι αυτοί που ήδη ανέφεραν ότι ο Σαλμάν εξέφραζε τη φωνή πολλών που μόνο του δεν μπορούσαν να αγωνιστούν να υψώσουν τη φωνή του. Και τι μειονότητε προστάτευε και καταπολεμούσε την αδικία. Ήθελε ένα δημοκρατικό καθεστώ. Και επέκρινε με δρυμή στόνου τον νόμο κατά τη βλασφημία. Ε, Εάν ο λαός μπορούσε να αποφασίσει, ο νόμο αυτός θα είχε ανακληθεί, θα είχε καταργηθεί. Όμως, ε, επίση ξέρουμε ότι έδωσε αγώνα για την ε, διάσωση μιας χριστιανής που είχε φυλακιστεί και είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Τελικά όλα αυτά του κόστησαν τη ζωή. Στήριξε όλες τις δυνάμεις του Πακιστάν που προσπαθούν να, να φέρουν την πρόοδο στη χώρα δεν είναι όλοι οι Πακιστανοί με το μέρος των ε, εξτρεμιστών. Άρα, στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και εμείς τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φίλε για να μας πει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, η συζήτηση αυτή είναι ακόμη μια απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλονίζεται από τέτοιε φρικτέ δολοφονίε όπω αυτή του κυρίου Τασίρ, του κυβερνήτη ε, του Πουντζάμπ στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Καπιστάν. Η Βαρόνια Άστον καταδικάζει την ε, αποτρόπια αυτή πράξη και παροτρύνει τι πακιστανικέ αρχέ να φέρουν του δράστε ενώπιον τη δικαιοσύνη. Η δολοφονία αυτή είναι τόσο περισσότερο θλιβερή καθώς βασίζεται στην προφανή και ρητή υπεράσπιση του κυρίου Τασίρ ε, υπέρ μιας χριστιανής που ήταν φυλακισμένη και κατά τις οποίες είχε ασκηθεί δίωξη. Ήδη το 2010 είχε εκφραστεί, είπατε, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Άστον, ε, κατά τη θανατική καταδίκη τη κυρία ε, Άζια Είχε ζητήσει από το Πακιστάν να καταργήσει την θανατική ποινή και να ε, σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα όπω τα ορίζουν οι διεθνεί συμβάσει τι οποίε έχει προσχωρήσει η χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένω έχει κάνει έκκληση για την ε, κατάργηση του νόμου κατά της βλασφημίας ε, στην ε, κυβέρνηση του Πακιστάν. Στα πλαίσια του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακιστάν ήδη έχει επισημανθεί ότι ο νόμος κατά της βλασφημίας ως έχει μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις και άσκηση πίεσης κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων. Γνωρίζουμε ότι οι ψευδείς κατηγορίες έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως ως εργαλείο για να επιληθούν ιδιωτικές διαφορές μεταξύ των πολιτών δηλαδή της χώρας αυτής και για προσωπικά κέρδη. Έχουμε δει βέβαια να κάνει κάποια βήματα η κυβέρνηση του Πακιστάν προκειμένου να προσπαθήσει να ε, διορθώσει κάποια από τα πιο αμφιλεγόμενα μέρη του νόμου. Ιδανικώ ε, ο νόμο αυτό θα πρέπει βεβαίω να, να, καταργηθεί πλήρω. Όμω ε, η περίπτωση αυτή τη δολοφονία του κ. Τασί δεν είναι η μόνη ατυχή περίπτωση. Υπήρξε και δημόσια στήριξη προ τον δολοφόνο. Αυτό μα ανησυχεί. διότι ε, είχε επικηρυχθεί όχι μόνο ο κύριος Στασίρα από τους εξτρεμιστές, αλλά και από άλλες δημόσιες προσωπικότητες που είχαν εκβαστεί κατά του νόμου ε, της βλασφημίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα βία και την ατιμορρησία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να τη δεχόμαστε. Η κυβέρνηση του Πακιστάν έχει την ευθύνη να προστατεύει τους πολίτες της. Και υπολογίζουμε στους υπευθύνους της κυβέρνησης ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών. Η δολοφονία του κυρίου Τασίρ ε, δείχνει ότι υπάρχει άνοδος και ε, επίταση του εξτρεμισμού στο Πακιστάν. Θα πρέπει όλα αυτά να τα σκεφτούμε, να δούμε ποιες θα είναι οι δικές μας αντιδράσεις, γνωρίζοντας σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή η κυβέρνηση και οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας έχουν ε, δραματικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουν. Εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Δεν υπάρχει ανελακτική παρά να εξακολουθήσουμε να ζητούμε την ενίσχυση των προοδευτικών δυνάμεων στο Πακιστάν και στην κοινωνία των πολιτών της χώρας αυτής. Το Σύνταγμα του Πακιστάν ρητό ε, διασφαλίζει την προστασία των ε, μειονοτήτων. Η κυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον εξτρεμισμό και όχι μόνο στι περιοχέ των σύνορων της την παραμεθόριο, αλλά και στου δρόμου των πόλεων του Πακιστάν. Θα πρέπει να, να, δώσουμε να δίνουμε διαρκή έμφαση στην, έμφαση... στην ε, εκπαίδευση συγγνώμη, και την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Και θα πρέπει να γίνουν περισσότερε προσπάθειε για να προωθηθεί η έννοια τη ανοχή στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, η ανοχή προ τι θρησκευτικέ μειονότητε. Όλοι γνωρίζουμε καλά πόσο ευάλωτη την κατάσταση κάποιων ε, πολιτών στο Πακιστάν λόγω των θρησκευτικών του πεπιθήσεων. Επειδή αποτελούν μέρη μειονότητα. Όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και οι Ινδουιστέ, η ΣΥΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να στηρίξει την προστασία τους και να μην επικεντρωθεί σε μία ομάδα ή θρησκευτικό δόγμα. Αυτό θα αποτελέσει όπλο στα χέρια όσων θέλουν να βαθύνουν τις διαφορές μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, δίνουμε προσοχή στην πλήρη προστασία όλων των ε, προσωπικών δικαιωμάτων, την ελευθερία της, ε, της, της των θρησκευτικών επιθήσεων στο Πακιστάν και παντού. Thank Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Έχει λήξει η συζήτηση για το θέμα του Πακιστάν. Έχω επτά προτάσεις ψηφισμάτων και θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία όταν ολοκληρώσουμε τις άλλες δύο